Πάμε στο επόμενο σημείο. Οι μονόλεπτες παρεμβάσεις, άρθρο 150. Ο κύριος Μότι. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί. Σήμερα 5 Μαΐου στην Ιταλία είναι η μέρα κατά της παιδοφιλίας και της παιδοπορνογραφίας. Πρόκειται για μία στιγμή σκέψης ε, όπως θεσπίστηκε από τον περσινό νόμο 41 για ένα φαινόμενο που είναι το οποίο διαδίδεται συνεχώς περισσότερο διότι σήμερα παιδόφιλος δεν είναι, αυτός που... δεν είναι ο γέρος που τσιμπάει το παιδάκι στο πάρκο αλλά είναι οργανωμένα κυκλώματα σε διεθνές επίπεδο και χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες όπως το ίντερνετ. Έτσι λοιπόν τα παιδάκια δεν είναι πια ήσυχα ούτε καν μέσα στα σπίτια τους. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφιερώσει και αυτή μία μέρα για αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό λοιπόν και έγραψα εγώ μία γραπτή δήλωση, ούτως ώστε να υπάρξει ένα γρήγορο σύστημα συναγερμού για να μπορούν να συνεργάζονται οργανωμένα οι αστυνομίες των κρατών μελών και να ανταλλάσσουν γρήγορα πληροφορίες. Εύχομαι αυτή η πρωτοβουλία να τύχει τη συμφωνία όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Μότι. Ο κύριος Μάτο. Την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρώπη έχασε μία μεγάλη ευκαιρία να απολευθερώσει την παγκόσμια αστροφυσική έρευνα για τα επόμενα 20 χρόνια. Αποφασίστηκε με αδιαφανείς διαδικασίες η Διεθνής Αστροφυσική Εταιρεία να εγκαταστήσει αυτό το τεράστιο τηλεσκόπιο στη Χιλή και όχι στην Ευρώπη. Αναρωτιέμαι όμως στην Ευρώπη κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Μία ευρωπαϊκή εγκατάσταση, ένα ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο το οποίο φτιάχτηκε με ευρωπαϊκά λεφτά να πάει να το στηθεί στην Ευρώπη, στην Αμερική εντός στην Ευρώπη. Τι έκανα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο έκανε τίποτα για να παρέμβουν τα κράτη-μέλη υπέρ της ευρωπαϊκής ε, υποψηφιότητας. Διότι στην Πάλμα των Καναρίων ίσως στη Λασπάλμας έπρεπε να πάει το τηλεσκόπιο. Και οι πολίτες της Λασπάλμας και οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πρόβλημα και θέλουν να ρωτήσουν γιατί. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πρότεινω ένα ψήφισμα για να σταματήσει η χρήση του κιανίου στα ανθρακοριχεία. Πρέπει να λάβουμε όλα τα μέτρα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και το περιβάλλον από οικολογικές καταστροφές. Ε, να, πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα σε όλο τον κόσμο για την προστασία του περιβάλλοντος. Και άμα θέλουμε να είμαστε παράδειγμα, γιατί δεν καταργούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την ουσία. Στο Μπαγιαμάρε πριν από 10 χρόνια έγινε ένα δυστύχημα με κιάνιο χειρότερο από το Τσερνομπίλ διότι κόσμος και κοσμάκι σε χιλιόμετρα και χιλιόμετρα επλήγει από αυτή την καταστροφή. Εγώ σήμερα Ευχαριστώ για την κατάργηση του, κανί, διότι πρέπει να σταματήσουμε να μολύνουμε τις ευρωπαϊκές περιοχές. Ο κύριος Μπουσόη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ελλάδα περνάει άσχημες ώρες. Αλλά και άλλες χώρες και άλλες χώρες περνάνε άσχημες ώρες και αποδεικνύεται ότι η οικονομική ρίση δεν έχει ξεπεραστεί, ότι υπάρχει πάντοτε ρίσκο για μεγάλη ανισορροπία. Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν μείωση των εισόδων τους, των δημοσιονομικών εσόδων και αυξάνουν τους φόρους. Αυτό συμβαίνει στη Ρουμανία. Η κυβέρνηση θέλει να αυξήσει τον ΦΠΑ και το φόρο των επιχειρήσεων. Αλλά μέσο πρόθεσμα και πρόθεσμα είναι καταστροφικά αυτά τα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρνει να διαμορφώσει μια κοινή στρατηγική για την οικονομική κρίση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών που έχουν λάβει μέτρα διαφορετικά μεταξύ τους. Και η μέθοδος αύξησης του φόρου δεν κάνει τίποτα παρά να εντείνει την κρίση. Ο Μπουρτσόφσκι δεν είναι εδώ. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους κερδοσκόπους οι οποίοι πλήττουν τις πιο ευάλωτες περιοχές του ευρώ. Μιλάμε για απώλεια εκατομμυρίων ε, ευρώ και δυστυχώς αυτό είναι πολύ μεγάλο ε, πλήγμα και έχει πολύ μεγάλη σημασία για τις ε, περιφερειακές οικονομίες. Μιλάμε ε, για μία ΕΚΤ η οποία υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητη αλλά δεν είναι. Υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο και την, τον ξέφρενο ανταγωνισμό του παγκοσμίου ε, κερδοσκοπικού κόσμου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταδείξουμε ε, αλληλεγγύη ως Ευρωπαίοι και να πληρώσουν αυτοί που πρέπει το κόστος αυτής της κλοπής. Εμείς δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε το μεγάλο μας αγώνα στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και θα θέλαμε να τιμήσουμε τους Έλληνες για το μεγάλο τους θάρρος. Ο κύριος Κόλμαν. Thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα την τραγική αυτή ημέρα κατέστη σαφές πως θα επιβληθούν δρακόν, μέτρα δρακόντιας λιτότητας στην Ελλάδα για να διαφυλαχτεί το ευρώ. Και όμως έτσι τιμωρείται ο ελληνικός λαός για το ότι ήταν σπάταλη η πολιτική του και για να διατηρηθεί η νομισματική ένωση. Εμείς θυμόμαστε το Σεπτέμβριο του 1992 στο Ηνωμένο Βασίλειο ή όπως λεγόταν τότε ο μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο μηχανισμός αιώνια ύφεση και τα καταφέραμε. Και όμως πραγματικά η λιτότητα λειτουργεί. Πρέπει λοιπόν να απελευθερωθούν οι Έλληνες από τα δεσμά του ευρώ, να κάνει το δούνο του τη δουλειά του και θα δείτε πόσο γρήγορα θα ανακάμψει η Ελλάδα όταν, όπως κάναμε και εμεί στο Ηνωμένο όταν φύγαμε από το μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμίων. Μην πληρώσει η Ελλάδα το τίμημα ενός ευρωπαϊκού υπερκράτους. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο για ένα λεπτό έχει κυρία Σήμερα παίρνω τον λόγο για την ασφάλεια των πτήσεων, το οποίο μας απασχόλησε πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Η ανθρώπινη ζωή είναι ένα αγαθό το οποίο είναι υπέρτερο οποιοδήποτε οικονομικού αγαθού Γι' αυτό ακριβώς η απαγόρευση των ε, πτήσεων ήταν απαραίτητη όταν είχαμε αυτό τον εξωτερικό κίνδυνο, δηλαδή την φυστιακή τέφρα. Υπενθυμίζω εδώ πέρα τις δύο καταστροφές που γλιτώσαμε παραλίγο το 82 και το 89 αλλά και τώρα όταν βρέθηκαν σε κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών υπολείμματα της ε, τέφρας. Γίνονται δοκιμές όταν οι ειδικοί δεν μπορούν να δώσουν οριστική απάντηση παραμένει γεγονός πως δεν θα πρέπει να ρισκάρουμε ανθρώπινες ζωές και θα πρέπει επίσης να δούμε ποιες είναι και οι εναλλακτικέ που έχουμε όταν δεν πετούν το αεροπλάνο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Λαντσίλα. Κύριε Πρόεδρε, Θεωρώ ότι για να βελτιωθεί η τροφιμική αλυσίδα στην Ευρώπη και να έχουμε μία καλύτερη διαφάνεια χρειαζόμαστε ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο να την Ευρώπη. Πρέπει οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ προμηθευτών και διανομέων να γίνουν καλύτερες. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε και τις πρακτικές κατά το του ανταγωνισμού. Οι νόμοι θα πρέπει να ερμηνεύονται κατά τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να βελτιώσουμε τους κανόνες ανταγωνισμού για να έχουμε μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ ΚΑΠ και εμπορικών πολιτικών. Αυτό είναι απαραίτητο για τις τιμές. Ο κύριος Σας ευχαριστώ. Εδώ συχνά κάνουμε λόγο για τη διακριτική μεταχείριση που υφίσταται η πολωνική μειονότητα στην Λιθουανία που δεν μπορούν να γράψουν καν το όνομά τους τα πολωνικά, κλείνουν τα πολωνικά σχολεία εκεί πέρα. Δεν επιστρέφεται η περιουσία τους μόνο και μόνο γιατί ήταν Πολωνοί η δε Επιτροπή Ηθικής της ε, ε, τιμώνησε τον κύριο Τόμασεύσκι όταν ρώτησε τον κύριο Μπαρόσο τι γίνεται με την πολωνική ε, μειονότητα. Και συνεχίζεται το σκάνδαλο στην, ε, στη Λιθουανία καθώς ε, τιμωρήθηκε εκεί πέρα ο υπεύθυνο ε, της ε, Πολωνικής Ένωσης γιατί έβγαλε φυλάδια σε δύο γλώσσες. Δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να τελειώσει αυτό το σκάνδαλο και να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ κύριε Καλινόφσκι. Τον λόγο έχει η κυρία Κάστεξ για ένα λεπτό. Δεν είναι εδώ η κυρία Κάστεξ. Η κυρία Σαβισάρ. Ούτε και αυτή είναι εδώ. Για να δούμε αν έχουμε τύχη. Ο κύριος Αγκουράκης Έχετε τύχει κύριε Πρόεδρε, είμαι εδώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, εκατομμύρια εργαζόμενοι απήργησαν και διαδήλωσαν σήμερα με το ΠΑΜΕ ενάντια στα βάρβαρα μέτρα που επέβαλε το κεφάλαιο η ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δούνο του. Τα μέτρα αυτά δεν είναι ούτε καινούρια και ούτε προσωρινά. Αποτελούν βάναυση εφαρμογή της καπιταλιστικής ανάπτυξης που οδηγεί σε κρίση και σε νέα κρίση αποσκοπούν στη διασφάλιση των κερδών της ελληνικής και ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας και στη συνέχιση της εφαρμογής της συνθήκης του μάστριχτ. εμπεριέχονται στη στρατηγική της λισαβόνας και της ευρώπης 2020. γι' αυτό είναι και αδιέξοδα. εμείς όμως λέμε ότι υπάρχει λύση. δεν είναι μονόδρομος η πορεία αυτή. είναι η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και μια ανάπτυξη με γνώμονα τις ανάγκες αυτών που παράγουν τον πλούτο. είναι η κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων και η λαϊκή εξουσία αυτή η πορεία ούτε οι προβοκάτσιες και ούτε οι εκβιασμοί της ελληνικής κυβέρνησης μπορούν να του σταματήσουν και ούτε τέτοιες δολοφονικές πράξεις σαν για αυτές που σημειώθηκαν σήμερα στην Αθήνα και μας συνταράσσουν όλους. Πιστεύουμε ότι η πορεία των ε, αγώνων του ελληνικού λαού θα είναι νικηφόρα. Ευχαριστώ κύριε Η πριν από λίγες ώρες θα λέγαμε πως ε, παρά την βεβήλωση ε, πολιτιστικών ε, μνημείων και την επανάληψη διαφόρων στερεοτύπων δεν αντιλαμβάνονταν το Συμβούλιο, την ελληνική κρίση ως ευρωπαϊκό ζήτημα, ούτε και η Κομισιόν. Αλλά λέγαμε πως οι Έλληνες θα υποστήριζαν την σοσιαλιστική τους κυβέρνηση στον αγώνα της για ανάκαμψη. Τώρα, υπό το βάρος των τραγικών γεγονότων των τελευταίων ωρών στην Αθήνα που πέθαναν τρεις άνθρωποι λόγω της βίας που προέκυψε από τα σκληρά οικονομικά μέτρα, υπενθυμίζω τα πρόσφατα λόγια του Ράσμουσεν. Η υποβάθμιση των ελληνικών ομολόγων σε τζάνκ είναι ενδεικτική της πολιτικής που ακολουθείτε. Νομίζω πως είναι επίγον για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ενισχύσουν τον αγώνα τους για την συνοχή. Ελπίζω αυτό το οποίο συνέβη πριν από λίγες ώρες στην Ελλάδα να μην είναι μεταδοτικό να μην μεταδοθεί κι αλλού και να σημειώσει αντιθέτως την αρχή μιας ομόφωνης προσπάθειας για σχηματισμό ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της αλληλεγγύης και της εταιρικής σχέσης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και πολύ ο Πρόεδρος. Η κυρία Όπως ξέρετε, εδώ και 120 χρόνια γιορτάζουμε την 1η Μαΐου. Είναι η μέρα του εργαζόμενου, η μέρα του εργάτη, η χειραφέτηση του εργάτη, έτσι ώστε η εργασία να μην αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης. 120 χρόνια μεγάλης ε, προόδου αλλά και παλινοδιών πότε αυτά τα καθολικά λόγια θα εισακουστούν έτσι ώστε να μην χάνονται ζωές και να μην γίνονται τόσο μεγάλες θυσίες. Δυστυχώς οι λαοί γνωρίζουν οπισθοδρομήσεις και παλινοδίες έτσι ώστε το μεγάλο κεφάλαιο να επιτίθεται. Όπως βλέπουμε στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και σε πολλές άλλες χώρες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτές, αυτή τη μάχη και να μην υπάρχει επιδείνωση της εκμετάλλευσης. Θα πρέπει να τιμούμε τους εργαζόμενους. Ο κύριος Θέλω να ευστήσω την προσοχή σας σε κάτι επίγον. Ένας ε, νεαρός Ιρλανδός, ο Μάικλ Ντουάερ, δολοφονήθηκε στην Βολιβία πριν από ένα έτος. Πολλοί πιστεύουν, πυροβολήθηκε και πέθανε, πολλοί πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε. Και είναι συγγενείς του παρόντες εδώ απόψε. Η μόνη επίσημη εξήγηση είναι πως ε, πέθανε σε απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου της Βολιβίας, κάτι το οποίο ε, μάλλον δεν ε, ισχύει αν σκεφτούμε τον χαρακτήρα του μάλλον ήταν μεμουμένος σε αυτή την προσπάθεια και δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις αρχές της Βολιβίας καθώς φαίνεται πως τα στοιχεία του ιατροδικαστή και της βαλιστικής εξέτασης είναι τελείως αντίθετα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από το Κοινοβούλιο και την κυρία Άστο να υποστηρίξει κυβέρνησης, τις προσπάθειες κυβέρνησης της Ισλανδίας για να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα αυτό το κάνουμε τη στήριξη των Ιρλανδών ε, Ευρωβουλευτών διακομματικά. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Η κυρία Γκόγκς. Ο κύριος Βίγενιν. Налага се да ангажирам вашето внимание с национален проблем – σας ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να αναφέρω έθνε, εθνικό πρόβλημα. Η Βουλγαρία κυβερνείται από μια ανίκανη λαϊκιστική κυβέρνηση που χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά του 1930. Ε, οι πιο λαϊκιστές είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Πρωθυπουργό. Εκατοντάδες ε, δημόσιοι υπάλληλοι που πρόσκειτο στην αντιπολίτευση απολύθηκαν. Είχαμε κτηνώδεις συλλήψεις πολιτών με παράλογες κατηγορίες. Οι δε πολιτικοί έδαιναν οδηγίες στην δικαιοσύνη και υπάρχουν σχέδια σύστασης ειδικού δικαστηρίου που θα λέγεται εξειδικευμένο δικαστήριο. Για πολλά χρόνια ζητούσατε από τη Βουλγαρία να κάνει περισσότερε προσπάθειε καταπολέμηση του εγκλήματο. Προσπάθειε γίνονται, αλλά φαίνεται πω καταπολεμείται η δημοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ευαίσθητο σε ζητήματα παραβίαση των δημοκρατικών αρχών. Θα έπρεπε να δείξει την ίδια ευαισθησία όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα σε κανένα κράτο μέλο. Σα ευχαριστώ, ο κ. Ζέγκερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. οικονομική κρίση, η ανεργία, η αύξηση του δημοσίου χρέους είναι οι βασικές προκλήσεις για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Να επιστήσω την προσοχή σας για κάτι το οποίο αφορά στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, την Ουγγαρία. Η ίδια φθορά δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να χειροτερεύει την κατάσταση και αυξάνει το δημόσιο χρέος. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση όθησε την Ουγγαρία σε άσχημη κατάσταση. Είτε για τους αυτοκινητοδρόμους, για τις επιχειρήσεις ή για ευρωπαϊκά σχέδια. Όλα όσα έγιναν σε αυτούς τους τομείς ήταν καθαρή διαφθορά. Και η διαφθορά παραμένει και σε περίοδο κρίσης. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να σταματήσει αυτό. Ο κύριος Μύρσκι. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιορτάζουμε την ε, νίκη κατά του φασισμού. Εν τω μεταξύ, 16 Μαρτίου, βετεράνοι των Waffen SS παρήλασαν ε, στο κέντρο της ε, Ρήγας. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουμε μπορέσει να σταματήσουμε αυτές τις ε, εκδηλώσεις. Η Ευρώπη, εν τω μεταξύ, συνεχίζει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. πάνω από 150.000 ε, ε, άνθρωποι, Ρώσοι, Ουκρανοί, σκοτώθηκαν από αυτούς τους ανθρώπους. Και όμως στη Λετωνία τους θεωρούν ε, ήρωες. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ κύριε Μίρσκι για ένα λεπτό ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ιστορία μας έδειξε πως από την κρίση μπορεί να οδηγηθούμε στην πρόοδο, από την πίεση να προκύψουν νέες ιδέες και ενωτόμοι μηχανισμοί για να οδηγηθούμε σε ανάπτυξη και να βγούμε από την κρίση. Θα ήθελα να τονίσω δύο τέτοιες ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν σε σωστά μέσα. Αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει σημασία, ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αξιολόγησης πρέπει να δημιουργηθούν. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που απαιτούνται, είναι κάτι που αξίζει τον κόπο εάν σκεφτούμε το μακροπρόθεσμα συμφέρον μας γιατί οπωσδήποτε θα έχουμε και άλλες κρίσεις στο μέλλον. Η ευρωπαϊκή κοινωνική οικονομία της αγοράς και το κοινό μας νόμισμα είναι βεβαίως θεμέλια του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και βεβαίως εάν έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο θα επιβληθεί έτσι το σύμφωνο σταθερότητα και θα έχουμε και ευρωπαϊκέ αξιολογήσει των οικονομιών. Πρέπει να τα συζητήσουμε σοβαρά αυτά και κατά την άποψή μου, καλό είναι να τα υιοθετήσουμε. Eh, Tiene la palabra. Έλεγα ευχαριστώ κύριε Γουίνκλερ και όχι κύριε Μίσκι. Ο κύριος Κρήτον έχει το λόγο. Asistăm în ultima perioadă la o ascensiune îngrijorătoare a extremei drepte și la radicalizarea. Ε, εμείς έχουμε μια άδικη άνοδο της άκρας δεξιάς μετά από τις εκλογές στην Ουγγαρία είδαμε ότι τα εξτρεμιστικά κινήματα έχουν ούριο άνεμο. Δεν αγαπούν ούτε τα γειτονικά κράτη, ούτε τις μειονότητες, ούτε την Ευρώπη. Εγώ διαμαρτύρομαι για όλα τα αρνητικά μηνύματα κατά των Ευρωπαίων πολιτών. Μία γαλλική τηλεόραση υβρίζει τακτικά τους Ρουμάνους. Και στη Βαρκελόνη υπάρχει και ένα πολιτικό κίνημα που είχε ως σύνθημα «Δεν θέλουμε Ρουμάνους εδώ». Ζητώ από <laughs> τις αρμόδιες αρχές να καταβάλουν προσπάθειες για να καταπολεμήσουν αυτό το επικίνδυνο φαινόμενο. Ο κύριος Αρσένης. πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συλληπιθώ τι οικογένειε των θυμάτων των σημερινών επιθέσεων στην αθήνα. αγαπητοί συνάδελφοι στο θέμα μα όμω θα είναι η κλιματική αλλαγή. οι 35.000 εκπρόσωποι των ηθαγενών πληθυσμών όλου του κόσμου που συναντήθηκαν στην κοτσαμπάμπα τη βολιβία μα θέτουν το δάχτυλο επί το τύπο των ήλων. μα ζητάνε να δεσμευτούμε στη συνδιάσκεψη του μεξικού για νομικά, με νομικό δεσμευτικά τρόπο για τη μείωση των εκπομπών μα. έχουν δίκιο δεν μπορούμε να αναβάλουμε πλέον αυτή την απόφαση. η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει άμεσα να δεσμευτεί επίσημα για μείωση 30% των εκπομπών στο 2020. αυτό θα αλλάξει τη δυναμική στι διαπραγματεύσει που είναι αλήθεια ότι έχουν πλέον κολλήσει με κίνδυνο να βληθεί η απόφαση για μείωση των εκπομπών για μετά το μεξικό και χωρί συγκεκριμένη ημερομηνία χωρί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και στο Κοινοβούλιο μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. 30% μείωση του αποτυπώματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 2020 έχει ήδη αποφασιστεί πρέπει να δείξουμε τον δρόμο στα κράτη μέλη μειώνοντας το αποτύπωμά μας κατά. 50%. όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στον καθημερινό χώρο εργασία μα και τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και μπορούμε και έχουμε υποχρέωση να την καταφέρουμε. Ευχαριστώ κύριε Αρσένη. Η κυρία Parlament το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα απαλλαγή στην ε, Κομισιόν και δικαίως γιατί ποτέ δεν είχαμε τόσο χαμηλό περιθώριο σφάλματος και βεβαίως ε, μόνο ο τομέας της ε, συνοχής ε, έχει ακόμα σημαντικό ποσοστό ασφαλμάτων, δηλαδή άνω του 5%. Επίσης θα πρέπει να δούμε ιδιαίτερα την γεωργία όπου έχουμε ένα ποσοστό ασφαλμάτων κάτω από το 2%. Οπότε λειτουργεί το σύστημα ελέγχου. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ και αυτά τα οποία αναφέρονται στην απαλλαγή για την Τουρκία, την προενταξιακή βοήθεια καθώς εκεί πέρα δεν υπάρχουν μετρήσιμα κριτήρια. Δεν είναι δυνατόν χωρίς μετρήσιμους δείκτες να πηγαίνουν χρήματα σε τρίτες χώρες. Ένας άμεσος έλεγχος των πληρωμών πρέπει να υπάρξει μόνο έτσι θα έχουμε άλλωστε και αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μορβάη έχει τον λόγο. Eh, ευχαριστώ. Το 11ο άρθρο της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπει ένα συγκεκριμένο δικαίωμα το οποίο όμως στην Ουγγαρία καταπατείται. Το Ουγγρικό στρατοδικείο καταδίκασε έναν συνδικαλιστή για μία δραστηριότητα που είχε να κάνει με την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και αυτό δεν συνέβη στον τρίτο κόσμο, αλλά σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύθηκε η στράτευση της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν αυτή την υπόθεση να τη θεωρήσουμε ως ένα πείραμα για να επαληθεύσουμε του λόγου το αληθος, Το αληθές. Και να δούμε πώς αυτή η θαραλέα γυναίκα θα μπορέσει να βρει το δίκιο της. Ευχαριστώ κυρία Στάνγκλου. δεν είναι εδώ. Οπότε τον λόγο έχει ο κύριος Γκέρκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ε, Πολωνία γίνεται εμπόριο ανθρώπων υπό διάφορα προσχήματα. Υπάρχουν τελείως ε, περίεργα πράγματα όσον αφορά την ενοικίαση ακινήτων μαζί με τους ενοικιαστές που συνήθως είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν είχαν δικαίωμα αγοράς οπότε ανεβαίνει συνέχεια το ενίκιο και βρίσκονται στον δρόμο. Παραβιάζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειαζόμαστε καλύτερα νομικά μέσα έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοια σκάνδαλα στην ε, Πολωνία. Πρέπει να προστατευτούν καλύτερα οι ενοικιαστές και χρειάζεται και κρατική ενίσχυση για τα θύματα αυτής της ε, τακτικής. Κλείνει. Το γύρο ο κύριος, ο κύριος Στογιάννοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο για να καταγγείλω μία αδικία. Μην νομίζετε πως δεν φταίνε οι Έλληνες για αυτά τα οποία έγιναν στην Ελλάδα. Η οικονομική κρίση οφείλεται ότι έχουν 14, 15 και 16 μισθούς το χρόνο πράγματα άγνωστα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για πολλά χρόνια έλεγε ψέματα η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τώρα λόγω των ψεμάτων αυτών οι Ευρωπαίοι ηγέτες ψήφισαν να δώσουν 110 δισεκατομμύρια ανταμοιβή στην Ελλάδα, ενώ η Βουλγαρία και η Εσθονία, που ήταν πειθαρχημένες θα τιμωρηθούν και θα καθυστερήσει η είσοδος του στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, είναι ανάξιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το οποίο συμβαίνει. Τιμωρούμε δηλαδή α, αυτούς που δεν φταίνε. Πρέπει να φύγει η Ελλάδα από την Ευρωζώνη. Ε, σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση στην ε,